Okay. I'm being Mr. Osman is very short... Μου λένε ότι ο κύριος Οσμάν κοντεύει να φτάσει, οπότε να ξεκινήσουμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν υπάρχουν εμ, αιτήματα για αλλαγέ, θα έλεγα να την εγκρίνουμε. Ωραία. Δεν έχω ανακοινώσεις από την πλευρά του Πρόεδρου Οπότε μπορούμε να εγκρίνουμε τα πρακτικά της συνεδρίασης της 9ης Σεπτεμβρίου. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνονται τα πρακτικά. Οπότε περνάμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Ανταλλαγή απόψεων με τους βραβευθέντες με το, με το βραβείο Ζαχάροφ. Έχουμε την Λοράν Σαλέ από την Βενεζουέλα πολύ σύντομα στο, στην αίθουσα μαζί μας. Όχι. Τον Λοράν Σαλέ. Και πολύ σύντομα θα έρθει και ο κύριος Σαλή Οσμάν. Είναι η πρώτη ε, ευκαιρία που έχουμε ως Επιτροπή να σας αποτίσουμε φορό τιμής για την αφοσίωσή σας στην προάσπιση των ανθρωπινών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Χαίρομαι ιδιαίτερος που μπορείτε να είστε μαζί μας σήμερα και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχετε εκτίσει δύο μακροχρόνιες πίνες φυλάκισης σε πολύ σκληρές συνθήκες και απελευθερωθήκατε μόλις πριν από, αποφυλακιστήκατε μάλλον μόλις πριν από λίγους μήνες. Την περασμένη χρονιά και το Σουδάν και η Βενεζουέλα πέρασαν πολύ δύσκολες στιγμές και σήμερα έχουν να αντιμετωπίσουν μείζονο σημασία δυσκολίες και προκλήσεις. Στην αρχή της χρονιάς το Σουδάν γνώρισε μια λαϊκή εξέγερση και βίαιη ε, καταστολή, η οποία οδήγησε στην ε, ε, ανατροπή του καθεστώτος του Προέδρου Ομάρ. Τον Ιούλιο το, ο στρατός και ένα συνασπισμό τη αντιπολίτευση μαζί με τη διαμαρτυρία αποφάσισαν ε, να μοιραστούν την εξουσία για τρία χρόνια και να οργανώσουν εκλογέ για να διοργανωθεί μια κυβέρνηση με εκπροσώπου τη κοινωνία των πολιτών. Θα θέλαμε λοιπόν να πάυσουν οι εχθροπραξίε στο εσωτερικό τη χώρα και να δημιουργηθούν δημοκρατικοί θεσμοί, ένα εύρο στο κράτο δικαίου και να υπάρξει οικονομική ανάκαμψη αλλά βεβαίω προ σε αβέβαιο δρόμο όλα αυτά. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε ουσιαστικέ βελτιώσει στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε περιοχέ ε, με συγκρούσει όπω τον Ταρφούρ, τον Νότιο Κορτοφάν και ο Γαλάζιο Νείλο. Όσον αφορά το Σουδάν, Αυτά για, μάλλον για το Σουδάν. Αλλά και η Βενεζουέλα βρέθηκε στο επίκεντρο τη προσοχή του Ευρωκοινοβουλίου. Το θεσμικό μα όργανο ενέκρινε τουλάχιστον πέντε ψηφίσματα, το πιο πρόσφατο τον Ιούλιο φέτο. Στο ψήφισμα αυτό το Κοινοβούλιο καταγγέλει τις παραβιάσεις των, δυνάμεων, των διοκτικών δυνάμεων και την βία καταστολή από τις ε, αρχές. Ε, καταδικάζουμε την εξάσκηση της ε, αθέρετης κράτησης των πανεσιανιστηρίων και των εξοδικαστικών εκτελέσεων, όπως ε, ε, και επιβεβαιώνουμε τη στήριξή μας για την έρευνα του Διεθνούς Δικαστηρίου για να δει τι εγκλήματα διαπράχθηκαν από το καθεστώ τη Βενεζουέλα. Επίση, το Κοινοβούλιο καλεί το Συμβούλιο να προβλέψει κυρώσει για τι κρατικέ αρχέ σε σχέση με τι παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταστολή. Ξέρουμε ότι βάσει των διεθνών οργανισμών υπάρχουν πάνω από 7 εκατομμύρια ε, άνθρωποι στη Βενεζουέλα που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ 94% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο τη φτώχεια και 70% των παιδιών δεν φοιτούν σε σχολεία. Ε, να καλωσορίσω λοιπόν τον κύριο Οσμάν. Ε, είμαι βέβαιη ότι οι καλεσμένοι μας θα μοιραστούν μαζί μας την ε, ε, συνοπτική εικόνα, την σφαιρική εικόνα που έχουν για το θέμα αυτό και θα μας ενημερώσουν για το Σουδάν και τη Βενεζουέλα. Να δώσω το λόγο στον κύριο Σαλή Οσμάν. Σας ευχαριστώ κύριε Οσμάν που μπορείτε να μας δώσετε τη δική σας οπτική γωνία για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα σας. Χάσατε την αρχή της συνεδρίασης. Αλλά χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε στην υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σήμερα, αυτό έλεγα. Και θα έλεγα, εάν δεν σας πειράζει, 8 λεπτά για τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ που μου δίνετε αυτήν την ευκαιρία να πάρω το λόγο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για ένα βραβείο το οποίο με τιμά ιδιαίτερα. Το πήρα το 2007 και με καλέσατε να πάρω το λόγο εδώ ενώπιόν σας. Να απευθυνθώ στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένα όργανο που πραγματικά είναι αρμόδιο για θέματα αδικίας που συμβαίνουν παντού στον κόσμο, ιδιαίτερα όμως θα σας μιλήσω για το Σουδάν. Όταν πήρα το βραβείο Ζαχάροφ, σας υπενθυμίζω ότι το έλαβα στο όνομα εκατοντάδων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν υποφέρει όπως και εγώ. Η τελευταία μου κράτηση, που ήταν η τρίτη φορά που φυλακίστηκα μετά από 13 χρόνια, η πέμπτη μάλλον φορά που ε, βγήκα από τη φυλακή ήταν στις 11 Απριλίου του 2019. Αλλά και το 18 βρέθηκα στη φυλακή και είμαι πολύ ευτυχής και πραγματικά εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι μπορώ να βρεθώ εδώ και πρέπει να σας πω ότι το Κοινοβούλιο με ιδιαίτερη θέρμη με υποστήριξε στέλνοντας επιστολές στην κυβέρνησή μου κατά τη διάρκεια της ε, κράτησής μου στις φυλακές. Και τις πέντε φορές που φυλακίστηκα δεν μου απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Απλώς μου προσάπτουν κάθε φορά ότι περασπίζομαι εκατοντάδες, χιλιάδες ε, θύματα τα οποίων τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται. Και νομίζω ότι κάποιοι από εσά γνωρίζουν ότι από το 2003, όταν ξεκίνησε αυτή η ιδιότητα στον Ταρφούρ, πάνω από 4 εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους, τα σπίτια τους. Και πάνω από 600.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από βομβαρδισμούς ε, μέσω αεροπλάνων και ελικοπτέρων. Καταστράφηκαν πάνω από 15.000 χωριά στην περιοχή του Νταρφούρ. αποτρόπια εγκλήματα έλαβαν χώρα. Εγκλήματα πολέμου και αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Εγώ είμαι στόχος τα τελευταία 7 χρόνια γιατί προσπάθησα να ακουστεί η φωνή ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Σήμερα η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης ε, στην χώρα μας δεν υπάρχει. Και η ατιμορρησία είναι κάτι που δυστυχώς επικρατεί. Τα εγκλήματα αυτά, γιατί πρόκειται για εγκλήματα για γενοκτονία, δεν τιμωρούνται από την δικαιοσύνη. Η κατάσταση λοιπόν στο Νταρφούρ έχει ε, περιγραφεί από τις προσφυγές μας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και από τις 3 Ιουνίου και τη σφαγή μπροστά στο στρατιωτικό επιτελείο στη Χαρτούμ, όπου εκατοντάδες άνθρωποι οι οποίοι απλώς διαδήλωναν ειρηνικά δολοφονήθηκαν. Σας ζητούμε λοιπόν να μην ε, χαθεί αυτή η δυνατότητα να εισακουστούν αυτά τα οποία προσπαθούμε να πούμε για άλλη μια φορά, να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ε, ευκαιρία έτσι ώστε να υπάρξει μια ανεξάρτητη διεθνής διερευνητική επιτροπή η οποία να μπορέσει να διαλευκάνει αυτά τα αποτρόπαια εγκλήματα. Και ήδη από το Δεκέμβριο του 2018 με την πρόσφατη εξέγερση ο αριθμός των θυμάτων πολλαπλασιάστηκε. Σας ζητάμε λοιπόν πραγματικά να σταματήσει αυτή η ατιμορρησία και η κυβέρνηση της Χαρτούμ να αλλάξει στάση. Η Ευρώπη πάντα μας στήριξε, η Ευρώπη πάντα ήταν στο πλευρό μας, αλλά τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε η Ευρώπη να έχει αλλάξει η στάση προς την κυβέρνηση της ε, Χαρτούμ και η διαδικασία της Χαρτούμ ε, αυτή τη στιγμή δεν είναι ικανοποιητική. Θα ζητάμε λοιπόν να αλλάξετε στάση, σας ζητάμε να μην ακολουθείτε τις παραπλανητικές ε, πληροφορίες που ακούτε από την κυβέρνησή μας. Δεν πρόκειται για μια κυβέρνηση η οποία διοικείται και διευθύνεται από πολιτικούς. Πρόκειται για μια κυβέρνηση, ναι, μεταβατική μεν, αλλά μια κυβέρνηση η οποία καθοδηγείται και διευθύνεται από στρατιωτικούς. Και κάποιοι μάλιστα από αυτούς που σήμερα βρίσκονται σε αυτή τη μεταβατική κυβέρνηση είναι μέλη της προηγούμενης ε, στρατιωτικής επιτροπής που κατήφθηνε τη χώρα μας ο Υπουργός ε, Άμυνας, ο Υπουργός Εσωτερικών. Δεν έχει αρμοδιότητα. Και πραγματικά, αν κοιτάξει κανείς αυτά που συμβαίνουν σήμερα όσον αφορά τι μεταρρυθμίσεις στο Σύνταγμα και στην νομοθεσία δεν αντικατοπτρίζονται καθόλου οι πραγματικές ε, προσδοκίες και τα αιτήματα των τελευταίων 13 ετών. Σας παρακαλώ πολύ λοιπόν να μην ξεχάσετε, να μην αγνοήσετε τις νόμιμες διεκδικήσεις ε, του λαού μας πρέπει πραγματικά να συνεχίσουμε την πορεία μας προς τη δημοκρατία, προς την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, προς το σεβασμό του κράτους δικαίου. Και αυτοί οι οποίοι έχουν διαπράξει αυτά τα αποτρόπαια εγκλήματα θα πρέπει να τιμωρηθούν, να δικαστούν. Και, εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται να υπάρχει μια σωστή αξιολόγηση και σωστά σημεία αναφοράς ε, όταν μιλάμε για αυτή την μεταβατική κυβέρνηση και την ε, κρίνουμε. Υπάρχει επίσης και η λεγόμενη μεταβατική δικαιοσύνη. Επαναλαμβάνω όμως ότι ο Μαρμπασίρ, και θέλω εδώ να μας υποστηρίξετε, πρέπει να προσαχθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εμείς ε, συνεχίζουμε τις ε, εκστρατείες μας ε, ζητώντας σας να δείξετε αλληλεγγύη, να σταθείτε στο πλευρό μας και ζητάμε πραγματική δικαιοσύνη. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριο Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Λοράν Σαλή και μετά θα έχουμε και τη δυνατότητα να συζητήσουμε τα θέματα αυτά, συνάδελφοι, να ακούσουμε τον επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να είμαι κοντά σας. Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που είχε έρθει σε συνεδρίαση η δική σας η μητέρα μου ζητώντας να με απελευθερώσουν. Εγώ τότε ήμουνα σε ένα κελί στη Βενεζουέλα, δεν είχα δικαστεί, δεν είχα περάσει καν από ανάκριση, ε, δεν είχα δικαίωμα ε, υπεράσπισης και είχα περάσει πάνω από τέσσερα χρόνια περίπου ε, φυλακή. Με λένε Λορέν Σαλέ, είμαι η περασπιστής των ανθρώπων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γεννήθηκα στη Βενεζουέλα. Στη Βενεζουέλα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πολιτική σύραξη. Αυτό που έχουμε στη Βενεζουέλα είναι μια ανθρωπιστική κρίση μια κρίση ε, ασφάλειας και αυτό το οποίο συμβαίνει στη Βενεζουέλα δεν είναι ε, πρόβλημα πολιτικών που δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Αυτό που συμβαίνει στη Βενεζουέλα είναι ή μάλλον δεν είναι μια μάχη διαφορετικών ομάδων για να κατακτήσουν την εξουσία, αλλά είναι το οργανωμένο έγκλημα το οποίο έχει αναλάβει την πολιτική διακυβέρνηση της χώρας και έχει σε ομοιρία όλους τους κρατικούς θεσμούς και επιβάλλει τρομοκρατία σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Τρομοκρατία. Η συστηματική χρήση βασανιστήριων έτσι ώστε ο πληθυσμός να σκύψει το κεφάλι και να διατηρηθούν στην εξουσία ε, με ατιμορρησία και να κάνουν λαθρεμπόριο χρυσού, κοκαίνης, πετρελαίου, να εκβιάζουν. Είναι ένα πρόβλημα ασφάλειας. Αυτό που συμβαίνει στη Βενεζουέλα δεν είναι το ότι κάποιοι επαναστάτες με καλές ε, ε, προθέσεις έχουν παρεκτραπεί. Αυτό που συμβαίνει είναι 20 χρόνια υπό τρομοκρατικό καθεστώς. Πριν από 71 χρόνια υπεγράφει η Συμφωνία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πριν από 71 χρόνια. Και σήμερα συνεχίζουν να δολοφονούν ε, τους ανθρώπους που είναι υπέρ ε, των ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων και υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα και δεν τα έχουμε αντιμετωπίσει σήμερα. Η ανθρωπότητα προοδεύει. Η τεχνολογία χρησιμοποιείται για πολύ θετικά πράγματα, αλλά επίσης και για πολύ αρνητικά η τεχνολογία χρησιμοποιείται ως εργαλείο βασανιστήριων. Ε, τα καταπιεστικά συστήματα έχουν ε, εξυγχρονιστεί. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη βασανιστήριου που μπορούν να κοροϊδέψουν τα ε, πρότυπα ε, και τους ε, κανόνες που έχουμε στη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Έχουμε τα λευκά βασανιστήρια, τη στέρηση ύπνου, για παράδειγμα. Έχουμε μέρη στη Βενεζουέλα που σήμερα έχουν κλείσει ανθρώπους και τους βασανίζουν. Εγώ δεν είμαι εδώ για να μιλήσω υπέρ ε, των πολιτών της Βενεζουέλας, αλλά υπέρ Ευρωπαίων πολιτών που έχουν φυλακιστεί στη Βενεζουέλα. Ξέρατε εσείς πως υπάρχουν κρατούμενοι Ευρωπαίοι στη Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι εδώ και μιλώ μαζί σας. Και υπάρχουν άνθρωποι σε ομοιρία που βασανίζονται στη Βενεζουέλα και είναι παράλληλα και Ευρωπαίοι πολίτες. Και είναι Ευρωπαίοι πολίτες, επαναλαμβάνω. Ξέρω πως είμαστε στην άλλη άκρη του κόσμου. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Δεν μπορούμε μόνοι μας εμείς οι πολίτες της Βενεζουέλας να αλλάξουμε κάτι. Τι να κάνουμε, να πάρουμε τα όπλα. Δεν πρόκειται. Γιατί εμείς είμαστε βαθιά δημοκρατικά. Δημοκρατικός λαός και το γνωρίζει η χώρα μου και το εκμεταλλεύεται η εξουσία. Εγώ δεν ήρθα για να σας πω ποια είναι τα αριθμητικά στοιχεία, πόσοι κρατούμενοι είναι, ποιοι έχουν φυλακιστεί για τα πολιτικά τους πιστεύω, γιατί εσείς τα στοιχεία αυτά τα έχετε και μπορείτε απλώς να κλικάρετε το τηλέφωνό σας και να τα βρείτε. Η, Μισελ Μπατσελέ που είναι η ύπατη εκπρόσωπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα που δεν μπορείτε να την κατηγορήσετε ούτε ότι είναι καπιταλίστρια ούτε ότι είναι προ-Γιάνκη, μίλησε ξεκάθαρα για το τι συμβαίνει στην Βενεζουέλα και ήρθα να σας ρωτήσω όπως ρωτώ σε άλλα κοινοβούλια πόσους ακόμα νεκρούς θα θρυνήσουμε, πόσους ακόμα θανάτους, πόσους πολιτικούς κρατουμένους ακόμα χρειάζεστε. Πόσους ακόμα πρέπει να βασανίσουν για να τους δολοφονήσουν και για να τους πετάνε από ε, τα μπαλκόνια όπως έγινε πέρυσι με τον λοχαγό Πέρες. Πόσους ακόμα πρέπει να δολοφανήσουν χωρίς να έχουν περάσει από δικαστήριο. Ας μας πει η ανθρωπότης ολόκληρη πόσα ακόμα, ε, πόσους ακόμα νεκρούς θέλει να μετρήσουμε. Πόσα ακόμα παιδιά πρέπει να πεθάνουν από την πείνα στη Βενεζουέλα έτσι ώστε να κάνετε κάτι. Πολλά μπορούν να γίνουν. Εγώ είμαι εδώ γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σας μιλώ, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δούλεψε για να απελευθερωθώ. Είμαι εδώ μπροστά σας, γιατί οι κυρώσεις οι οποίες επιβλήθηκαν κατά των ε, υπαλλήλων ε, και των υψηλά ιστάμενων ε, υπαλλήλων του καθεστώτος, οι εξατομικευμένες κυρώσεις δεν είναι μόνο ένα πρακτικό τρόπο για να εφαρμόζεις τη διπλωματία, είναι ένας πραγματικά εξαιρετικός τρόπος να επιβάλλεις την ηθική και τους κανόνες. Γιατί αυτοί οι οποίοι παραβιάζουν συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα συνεχίζουν να ζουν χωρίς να τιμωρούνται. Γιατί ο μεγάλος κίνδυνος από όλα αυτά είναι το μήνυμα το οποίο στέλνουμε τους νέους όλου του κόσμου. Ποιο είναι το μήνυμα αυτό. Ότι μπορείς να εγκληματίσεις. Μπορείς να παραβιάσεις τον νόμο. Αρκεί να εξασφαλίσεις το εξή. Να είσαι αρκετά σκληρός, αρκετά διαστραμμένος. και να κάνεις κακό σε πάρα πολλούς, έτσι ώστε να μην τιμωρηθείς ποτέ. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουμε. Και όταν βλέπουμε τέτοιους δολοφόνους όπως ο Νίκολας Μαδούρο, όπως ο Καβέγιο και δεν τρέχει τίποτα, τότε τι λέμε στον κόσμο, ότι τους κοροϊδεύουν. Τους κοροϊδεύουν συνέχεια και τα παιδιά στη χώρα μου συνεχίζουν να πεθαίνουν από την πείνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που λάβατε υπόψη το τι συμβαίνει στη χώρα μου. Σας ευχαριστώ πολύ. για την κληρονομιά του Ζαχάροφ που εσείς υπερασπίζεστε και που για μας σημαίνει τόσο πολύ και αξίζει η δουλειά που κάνετε. Είναι πολλές οι προσδοκίες από τη δική σας επιτροπή και ελπίζω πως όπως είμαι εγώ ελεύθερος, όπως είναι ο Οσμάν ελεύθερος, έτσι θα βοηθήσετε και αυτούς που είναι στην Κούβα, στο Γουαντάναμο, στην Ικαράγουα, στη Σαουδική Αραβία θα απελευθερωθούν γιατί και αυτοί θύματα είναι. Και εσείς έχετε τη δύναμη να ανοίξετε, να σπάσετε τα λουκέτα. Γι' αυτό προσπαθήστε. Και εμείς θα βρεθούμε εκεί, θα σας στηρίξουμε και θα συνεργαστούμε μαζί σας για, μια, για ένα κόσμο ο οποίος θα είναι πιο ελεύθερος και πιο δίκαιος. Σας ευχαριστώ. Thank Ευχαριστούμε πολύ και τους δυο σας για αυτές τις μαρτυρίες. Εγώ ως νέο μέλος του Κοινοβουλίου θεωρώ ότι αυτά τα μηνύματα, αυτές οι μαρτυρίες δείχνουν πόσο σημαντικό είναι το βραβείο Ζαχάροφ και τι ε, μπορούμε εμείς να προσφέρουμε. Διότι το γεγονός ότι έχετε έρθει εσείς οι δύο εδώ σήμερα δείχνει ότι τα πράγματα ε, κάπως κινούνται και έχουμε κάτι κάνει. Ε, άρα χαίρομαι πολύ που είστε και οι δύο εδώ που και βρίσκεστε εδώ μαζί μας, αντί να βρίσκεστε σε ένα κελί στη φυλακή. Να δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους. Έχουμε περίπου μισή ώρα για την ανταλλαγή απόψεων. Να ξεκινήσουμε με την κυρία Φισλέρ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ που έχετε έρθει σήμερα. Κύριε Σαλή Οσμάν, κύριε Λοράν Σαλή, ευχαριστούμε για τις μαρτυρίες σας. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικές και ειλικρινά αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη. Χθε, κατά την ακρόαση του κυρίου Μπορέλ, που είναι ο ύπατος εκπρόσωπος ε, υποψήφιος τουλάχιστον, ε, αναφέραμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τώρα η Βενεζουέλα και συμφωνεί. Συμφωνεί ότι η κατάσταση ε, είναι πια ε, σε, ανθρωπιστικό επίπεδο ανησυχητική. 25 πολίτες της Βενεζουέλας ε, και είναι μέλη της κυβέρνησης, είναι σε κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή κυρώσεων. Σκοπεύουμε να αποδώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο τι ε, θα γίνει σχετικά και στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλουμε να δούμε τι δυσκολίες υπάρχουν λόγω της μετανάστευσης από την Βενεζουέλα προς την Κολομβία. Ήθελα να ρωτήσω, οι κυρώσεις που προβλέπονται αυτή τη στιγμή θεωρείτε ότι είναι αποτελεσματικές, δραστικές, πιστεύετε ότι χρειάζονται διαφορετικές, πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα και εν τέλει, βρίσκεται ότι ο διάλογος που γίνεται αυτή τη στιγμή μπορεί να αποφέρει καρπούς. Κύριε Ουσμάν, οι βίες καταστάσεις που περιγράφετε, δεν ξέρω και τι να πω, είναι δύσκολο να τη σχολιάσω και πραγματικά ανησυχώ για το τι περνάνε οι γυναίκες και τα παιδιά. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω. Και επίσης τι μπορούμε εμείς από την πλευρά μας ως ευρωβουλευτές να κάνουμε για να έχουμε μια θετική επίδραση, να αναχαιτήσουμε, να καταπραίνουμε αυτές τις καταστάσεις βίας. Πραγματικά χαίρομαι που το βραβείο Ζαχάροφ σας έχει απονεμηθεί και σας ευχαριστώ για όλα όσα κάνετε. Σας ευχαριστώ προσωπικά. Ευχαριστούμε κυρία Βισλέρ Λίμα. Θα έλεγα να ακούσουμε δύο ακόμα ερωτήσει και μετά να περάσουμε στο γύρο των απαντήσεων. Ε, η κυρία Σάντου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε και τους δυο σας που είστε εδώ και χαιρετίζω και τον Σαλή. Οι μαρτυρίες που μας δώσατε πραγματικά μας αφήνουν άφωνους. Δεν έχει κανείς λόγια. Να κόβουν την ανάσα. Είναι δραματικά τα γεγονότα, οι καταστάσει είναι πραγματικά πολύ βαριέ για θέματα παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για καταστάσεις βίας. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδιάφοροι ούτε ως πολιτικοί θύνοντες, ούτε ως ανθρώπινα όντα, όπως είμαστε όλοι μας. Και άκουσα τον ε, Σαλέ τη μαρτυρία του. Έχω παρακολουθήσει τον αγώνα του, τον αγώνα όλων στην Βενεζουέλα και η πορτογαλική κοινότητα στη Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή που είναι και πολυπληθής ζει σε ανθρωπιστικές συνθήκες ε, επισφαλής. Είναι μια κατάσταση που εμείς στην Πορτογαλία την ε, παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή και ανησυχία και, ανησυχία. και το βραβείο Ζαχάροφ κάπως βοήθησε ίσως να αλλάξετε κάτι στη ζωή σας. Βέβαια η κατάσταση στη χώρα σας δεν έχει οδηγηθεί σε λύση. Μιλήσαμε και για το θέμα των κυρώσεων και αυτό είναι κάτι που επανειλημμένως το έχουμε συζητήσει μεταξύ μας. Το συζητάμε διαμακρών και θα συνεχίσουμε να το συζητάμε και στο προσεχές μέλλον. Τι είδους όμως κυρώσεις και σε τι βαθμό θεωρείτε ότι μπορεί να είναι αποτελεσματικές. Ήθελα να μας μιλήσετε γι' αυτό και κυρίως θέλω να μας πείτε ποια είναι η δική σας η οπτική γωνία για το πώς θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε αυτό το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί στη Βενεζουέλα. Τι χρειάζεται να γίνει στην πράξη, τι χειροπιαστό χρειάζεται για να αλλάξει η κατάσταση και να υπάρξει μια ειρηνική λύση, μια οριστική λύση για την ε, κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Και ξέρω ότι πληροφορίες έχετε ε, από το τι συμβαίνει στη χώρα σας στην πράξη. Ποια είναι η δική σας η θεώρηση για αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες ως προς την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια. Ε, ανθρωπιστική βοήθεια που χορηγείται σε ποιε ομάδε του πληθυσμού δυσκολεύεται να φτάσει ή όχι. Γιατί εγώ έχω πολύ αντιφατικέ πληροφορίε. Ήθελα και αυτό, αν μπορείτε κάπω να το σχολιάσετε. Για τον κύριο Οσμάν, γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά την κατάσταση, την ε, πραγματικά θλιβερή κατάσταση που περνάει η χώρα σας. Είναι δραματικές οι συνθήκες, η βία είναι ανίποτη τα ακούμε από τους πρόσφυγες που χρήζουν διεθνούς προστασίας και φτάνουν τα πολλά σε ευρωπαϊκές χώρες. Οι μαρτυρίες τους είναι πραγματικά ε, δραματικές. Και το ίδιο ερώτημα που έθεσα και στον κύριο Σαλή θα θέσω και σε εσά. Ποια είναι η δική σας η οπτική γωνία, η προοπτική για την ε, ενδεχόμενη λύση της κρίσης στη χώρα σας και σε τι βαθμό εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε. Ποιες θα ήταν οι καταλληλότερες μέθοδοι για να επιτρέψουμε μια λύση σε όλη αυτή την κατάσταση. Και ως προς την ανθρωπιστική βοήθεια, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί και από τη δική σας χώρα οι πληροφορίες μας φτάνουν είναι αντιφατικές για τη χρήση αυτής της ανθρωπιστικής βοήθειας και το πώς φτάνει σε αυτούς που την έχουν περισσότερο ανάγκη. Γνωρίζουμε ότι Πραγματικά η βοήθεια, η ανθρωπιστική στη χώρα σας είναι άκρος αναγκαία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κυρία Σάντους. Κυρία Βόλαντα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Κύριε Σαλή, κύριε Οσμάν, σας ευχαριστώ για τις μαρτυρίες σας και όσα κάνετε για τα ανθρώπινα δικαιώματα ιδίω για το Σουδάν. Ξέρουμε ότι η τωρινή κυβέρνηση ε, προέκυψε ε, λόγω συμβαστική λύσης, μιας συμφωνίας. Όμως ο κύριος Χαμτάγκαλο από το 2019 φαίνεται να είναι συνυπεύθυνος για τις φαγές στο Χαρτούμ και εκπρόσωποι του στρατού ε, τώρα στο νέο συμβούλιο που κυβερνά τη χώρα έχουν έδρα ε, και θέση. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί που συμμετέχουν στις πολιτικές δομές και τι θα γίνει με τις ε, αυξανόμενες παραβιάσεις καθώς και τις εχθροπραξίες ή τη σφαγή στο χαρτούμ. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ώστε κάποια στιγμή στο μέλλον να υπάρξει ένας διάλογος να οργανωθεί κάτι και να δοθεί μια λύση στα όσα συνέβησαν στο παρελθόν. Και η ερώτησή μου προς τους δυο σας είναι το βραβείο Ζαχάροφ είχε κάποια διαφορά, έκανε κάποια διαφορά για το έργο σας. Μπόρεσε να σας δώσει μια όθηση για να προστατεύσετε καλύτερα τα ανθρώπινα δικαιώματα που προασπίζεστε. Είναι κάτι που μείωσε την πίεση η οποία ασκείται εναντίον σας. Και στο μέλλον μπορεί να διοργανωθεί κάποιος διάλογος, διότι ξέρουμε ότι η βασική, πρόθεση, η βασική προϋπόθεση για να υπάρξει μια θετική εξέλιξη στις υποθέσεις και των δύο χωρών σας είναι να μπορέσει να οργανωθεί κάποιο είδους διάλογος. Δώσω το λόγο στους ε, προσκεκλημένους μας, κύριε Σμάν, και κατόπιν άλλος ένας γύρος ερωτήσεων θα ακολουθήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ σημαντικές ε, οι ερωτήσεις όλων σας. Σας ευχαριστώ που ανησυχείτε και νοιάζεστε για μας. Τώρα, για την ερώτηση που αφορά τα παιδιά. Ήθελα να σας πω ότι μετά την τεράστια ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή του Δαρφουρ μετά την καταστροφή κοινοτήτων αυτό που συνέβη είναι ότι οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους στα σπίτια τους και να συγκεντρωθούν σε στρατόπεδα ειδικά για τους ε, εκτοπιστέντες. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όσον αφορά τη σύνθεση αυτών των ε, εσωτερικά εκτοπιστέντων ε, προσώπων, το 80% αυτών είναι γυναίκες και παιδιά. 80% αυτών που διαμένουν σε αυτά τα στρατόπεδα είναι παιδιά και γυναίκες. Οι άντρες είτε βρίσκονται σε μπόλεμες ομάδες, είτε έχουν χάσει τη ζωή τους, είτε αναγκαστικά εγκατέλειψαν την περιοχή του Νταρφούρ, είτε ακόμα και τη χώρα, εγκατέλειψαν το Σουδάν και έφτασαν ε, στην Ευρώπη, στις Ηνωμένε Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία. Κυρίως λοιπόν γυναίκες και παιδιά είναι ο πληθυσμός που παραμένει σε αυτά τα στρατόπεδα. Εγώ λοιπόν εξ ονόματος των ε, επιζώντων και των θυμάτων. Πιστεύω ότι η θέση της Ευρώπης ήταν καθοριστική για να μπορέσουν να επιβιώσουν όλα αυτά τα άτομα, χιλιάδες άνθρωποι, γιατί η ανθρωπιστική βοήθεια η οποία προέρχεται από τα ευρωπαϊκά κράτη είναι εξαιρετικά σημαντική. Και από τον Καναδά βεβαίως, την Ιαπωνία, Πρόκειται για χώρες που έχουν έμπρακτα δείξει την ε, αλληλεγγύη τους όλα αυτά τα χρόνια και βοήθησαν όλους αυτούς τους επιζώντες και τα θύματα να είναι ακόμα εν ζωή. Ο Μαρμπαζίρ βεβαίως, όπως ξέρετε, έχει πάρει την απόφαση να απελάσει όλους τους εκπροσώπους των ΜΚΟ και όλους αυτούς οι οποίοι εργάζονται και παρέχουν αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια. Τώρα, με τις γυναίκες. Εγώ εργαζόμουν σε μία μικιό που ήταν ε, δραστηριοποιημένη σε θέματα βασανιστήριων. Sudan Organization Against Torture και πρέπει να σας πω ότι αυτά που συνέβησαν ήταν φρικιαστικά και τα θύματα ήταν ε, γυναίκες και παιδιά. Υπάρχουν πολλές προσφυγές ε, στα δικαστήρια του Σουδάν. Όπως σας είπα όμως η δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη. Και αυτό που ακούμε πολλές φορές από τα θύματα είναι ότι όσο χρόνο και να πάρει αυτή η διαδικασία, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να ακουστούν αυτές οι μαρτυρίες, να γραφτούν τα ονόματα των θητών, αυτών που έχουν διαπράξει αυτά τα εγκλήματα, όσα χρόνια και να πάρει αυτή η διαδικασία. Και βεβαίως να υπάρξει λογοδοσία, να υπάρξει τιμωρία για αυτούς που έχουν διαπράξει αυτά τα εγκλήματα. Για πρώτη φορά πρέπει να σας πω ότι διαπιστώσαμε την τροπή των ε, νεαρών κοριτσιών και των γυναικών. Δεν ήθελαν να περιγράψουν αυτά τα εγκλήματα. Πολλές φορές βλέπουμε αυτά τα εγκλήματα να έχουν διαπραχθεί ενώπιον ανδρών της οικογένειας, των ε, πατεράδων τους, των ε, συζύγων τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά είχαν σε σκοπό τον εξευτελισμό, την ταπείνωση. Γι' αυτό και πλησιάσαμε σημαντικά πρόσωπα από τις κοινότητες τους, θρησκευτικού ηγέτες, οι οποίοι μπόρεσαν να πείσουν τα νέα κορίτσια και τις γυναίκες να μιλήσουν. Μιλήσαμε για εκατοντάδες χιλιάδες τέτοιες περιπτώσεις, αλλά ούτε μία από αυτές δεν έχει ε, δικαιώσει τα θύματα ενώπιον των δικαστηρίων του Σουδάν. Η ατιμορρησία λοιπόν συνεχίζεται. Αυτή είναι η κατάσταση. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν παρόλα αυτά κάποιες πολύ δυνατές θαραλές γυναίκες, οι οποίες πήραν το λόγο και περιέγραψαν την κατάσταση. Και θα επανέλθω εδώ στην ομιλία μου στο Κοινοβούλιο όταν είχα πει ότι συνεχίζουμε να έχουμε ελπίδα. Διότι έχουμε γυναίκες, αδερφές, μητέρες, ηλικιωμένες γυναίκες στα στρατόπεδα, οι οποίες μάχονται να διατηρήσουν ζωντανές τις κοινότητές μας, τη μνήμη και την ιστορία παρόλο που αυτό που τελικά προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση είναι εθνοκάθαρση. Και χιλιάδες, εκατομμύρια άτομα είναι εγκλωβισμένα στα στρατόπεδα αυτά και δεν τους επιτρέπεται να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Οι γυναίκες λοιπόν και τα παιδιά στα στρατόπεδα πραγματικά προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανές τις παραδόσεις μας, την ιστορία μας, τη μνήμη, για να μην πέσει σε λύθη όλη αυτή η ιστορία. Μιλούν στα παιδιά, μιλούν στις νεότερες γυναίκες. Αλλά πραγματικά ακόμα τους απαγορεύεται η επιστροφή στα χωριά τους και στα σπίτια τους και τους δίνονται κάποιες εναλλακτικές λύσεις. Αλλά πραγματικά πρόκειται ξεκάθαρα για μια προσπάθεια εθνοκάθαρσης. Αυτά είχα να πω. Και όσον αφορά τους πρόσφυγες, πάρα πολύ ανησυχητικό φαινόμενο. Εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους, δεν έχουν που να διαφύγουν, δεν είναι πουθενά ασφαλείς και ξέρετε ότι πολλές φορές νέοι έρχονται στην Ευρώπη μέσω, μέσω πολύ επίπονων όπως ξέρετε, διαδρομών φτάνουν στη Λιβύη, συλλαμβάνονται. Ξέρετε ότι στην Λιβύη υπάρχει εμπόριο προσφύγων. Ξέρετε τις συνθήκες ε, κράτησης και πώς τελικά περνάνε τη Μεσόγειο οι άνθρωποι αυτοί, ελπίζοντας ότι η Ευρώπη είναι ένας παράδεισος. Κάποιοι από αυτούς τους ε, πρόσφυγες όντως ε, παρουσιάζουν προβλήματα, είναι άτομα που έχουν ε, επαφές με την τρομοκρατία, έχουν φανατιστεί, ανήκουν σε ακραίες ε, θρησκευτικές οργανώσεις, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς υποφέρουν. Υποφέρουν και πρέπει να εγκαταλείψουν την χώρα τους για να σώσουν τη ζωή τους. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος, με ρωτάτε, να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Θα πρέπει να σταματήσει η κυβέρνηση αυτήν την εμπόλεμη κατάσταση στον Ταρφούρ και στις άλλες περιοχές που συνεχίζουν να μαστίζονται από τη βία. Θα πρέπει επίσης να μιλήσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε όλους για την ανάγκη να επανέλθει η δημοκρατία, να σταματήσει αυτή η ατιμορρησία, να πούμε όχι στη δικτατορία η Ευρωπαϊκή Ένωση με το ξεκίνημα της διαδικασίας της Χαρτούμ έχει σήμερα, αν θέλετε, αμαυρίσει την εικόνα της, διότι η συνεργασία με αυτήν την κυβέρνηση έχει δυστυχώς επιδεινώσει την εικόνα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί εδώ θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μην εθελοτυφλούμε. Πρόκειται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνεχίζονται. Πρέπει λοιπόν να ξανασκεφτείτε την στάση σας. Πρέπει να υπάρχει μια αξιολόγηση της κατάστασης, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ειρηνικό περιβάλλον. Και αυτή η μεταβατική κυβέρνηση θα πρέπει πάνω απ' όλα να κυρώσει τις πολύ σημαντικές διεθνείς συμβάσεις, παραδείγματος χάρη για την εξάλληψη των βασανιστήριων, για την εξάλληψη κάθε είδους διακρίσεων. Αυτά είναι βήματα που αποτελούν την προϋπόθεση για την οποιαδήποτε ε, συμφωνία που ενδεχομένως θα υπογραφεί με την κυβέρνηση αυτή. Η Ευρώπη λοιπόν θα πρέπει πραγματικά να κρατήσει την θέση της. Ας μιλήσουμε όμως και για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, στο οποίο θα πρέπει να προσαχθούν όλοι οι εγκληματίες. Και αυτό είναι πραγματικά επίγον. Τέλος, Θα ήθελα να μιλήσω για τους συμβιβασμούς. Οι συμβιβασμοί για την μεταβατική κυβέρνηση. Γιατί έγιναν αυτοί. Διότι υπήρξε μια εξωτερική παρέμβαση από μέρους της Αραβίας, της Αιγύπτου και με αυτόν τον τρόπο παρέμεινε στην εξουσία η παρούσα κυβέρνηση. Αλλά πρέπει και η Ευρώπη να πιέσει στο εσωτερικό της χώρας μας θα πρέπει να συνεχίσει η μετάβαση προς τη δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο. Bueno, la Η ανθρωπιστική βοήθεια. Όταν ένα παιδί ε, λιμοκτονεί, η βλάβη η οποία προκαλείται είναι μόνιμη και δεν είναι αντιστρέψιμη. Και αυτό είναι οδυνηρό για μας, γιατί ξέρουμε πως τα παιδιά αυτά τα οποία ε, λιμοκτονούν ή θα πεθάνουν ή θα έχουν προβλήματα σε όλους τη ζωή. Και αυτό δεν είναι λίγο. Θα είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Εμένα με τρομάζει το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας, γιατί τι γίνεται. Δεν λύνουμε το βασικό πρόβλημα και απλώς διαχειριζόμαστε κάποιες περιφερειακές διαστάσεις του προβλήματος. Αυτό δεν βοηθά στο να αλλάξουμε κάτι. Αντίθετα, μονο, μονιμοποιούμε κάποιες καταστάσεις. Αυτό που με ανησυχεί λοιπόν είναι το ότι συνηθίζουμε στο να μας τρέφουν από ξένες χώρες τα οποία έρχονται κυβότιο-κυβότιο από τα σύνορα και η ανθρωπότητα συνηθίζει στο να στέλνει τρόφιμα στη Βενεζουέλα. Γιατί αυτό δεν λύνει τίποτα. Καταρχήν δεν φτάνει καν σε ένα ποσοστό αντιπροσωπευτικό της κοινωνίας. Δεν φτάνει. Εγώ υποψιάζομαι πως στις χώρες όπου είχαμε ανθρωπιστικές κρίσεις τέτοιου είδους, τι γίνεται, δημιουργείται ένα οικονομικό και πολιτικό οικοσύστημα που βασίζεται στην ανθρωπιστική βοήθεια, που διατηρεί εν ζωή ε, την κρίση στο διηνικές. Η καλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια που μπορείτε να μας στείλετε είναι να ε, ε, διώξουμε τη δικτατορία, το να καταδικάσει η Ευρώπη τους υπέτειους για αυτά τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αυτή είναι η καλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια. Δηλαδή το γάλα, το τυρί, το κρέας που στέλνετε με την ανθρωπιστική βοήθεια και που χρειάζονται οι κάτοικοι της Βενεζουέλας είναι τα τρόφιμα τα οποία παράγουμε εμείς ήδη. Το δικό μας γάλα τυρί και κρέας. Γι' αυτό λοιπόν θα ε, πρέπει να καταπολεμήσουμε μια δικτατορία η οποία δεν επιτρέπει ε, στην χώρα μας ε, να τραφεί με δικές της δυνάμεις. Γιατί είναι στρατιωτικοί στην εξουσία και αυτοί ούτε καλλιεργούν ούτε αρμέγουν. Το μόνο που κάνουν είναι διαπραγματεύονται με εταιρείε στην Ευρώπη και στο Μεξικό για να αγοράσουν εκεί τρόφιμα και να πάρουν προμήθειες από τα χρήματα αυτά και ζουν από αυτέ τι προμήθειε και στη Βενεζουέλα για το λόγο αυτό κατέστρεψαν την παραγωγική οικονομία και μέσω τη πείνα ε, διατηρούν υποταγμένο τον πληθυσμό γιατί η πείνα για μια δικτατορία είναι πολιτικό εργαλείο. Γι' αυτό δεν πρόκειται όσο υπάρχει η δικτατορία αυτή να ξεπεράσουμε την πείνα γιατί ξέρετε πως κάποιος που έχει άδειο στο μάχη δεν σκέφτεται. Κάποιος που πεινάει υποτάσσεται. Υποτάσσεται μέχρι τέλους. Κάποιος που πεινάει δύσκολα θα δώσει τη μάχη πέρα των δικαιωμάτων του. Κυρώσεις. την πρώτη φορά που βγήκα να μιλήσω στον κόσμο για το τι συμβαίνει στη Βενεζουέλα και να ζητήσω βοήθεια ήταν το 2008. Και το 2018, ε, δέκα χρόνια μετά, με δέχτηκαν στην υπατιαρμοστία. Είδα λοιπόν όλες τις εξελίξεις στην διεθνή κοινότητα σε σχέση με τη δικτατορία στη χώρα μου. Η δικτατορία στη χώρα μου, όπως και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, δεν φτάνει σε τόσο σκληρές διαστάσεις αν δεν το επιτρέπει η διεθνής κοινότητα. Για μια δικτατορία να κάνει όλα αυτά που κάνει στη Βενεζουέλα χρειάστηκε και χρειάζεται μια διεθνή κοινότητα που αγοράζει από αυτήν και που τις πουλάει. Δηλαδή να αγοράζει πετρέλαιο και να πουλάει όπλα. Και αυτό για πολλά χρόνια. Αυτό συνέβαινε και χαμογελούσαν στον Όγκο Τσάβης και στην αρχή χαμογελούσαν και στον Μαδούρο. Οπότε μόνοι εμείς δεν μπορούμε αυτό να το αναστρέψουμε. Το είπες και εσύ, πού είναι η δικαιοσύνη, ποιο είναι το δικαστήριο. Τέσσερα χρόνια, ένα μήνα και επτές μέρες ήμουνα μέσα σε ένα κελί. Δυόμιση χρόνια ήμουνα σε ένα κελί κάτω από το έδαφος. Ήτανε σαν μαύρος τάφος και ακόμα δεν με έχουν δικάσει. Το, το Διεθνές Δικαστήριο χρωστά στην ανθρωπότητα. Θα πρέπει και αυτό να το αξιολογήσουμε. Γιατί το έχουμε στήσει. Και οι κυρώσεις είναι από τα λίγα όπλα που έχουμε στα χέρια μας. Εγώ προτιμώ να επιβάλλετε κυρώσεις και να καταστρέψετε ε, αυτές τους δεσμούς τους οικονομικούς που έχει η δικτατορία ε, ε, μέσω συναλλαγών παρά να μας στείλετε ένα αεροπλάνο με, να βομβαρδίσει. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί ε, μία, έναν αυτοκινητόδρομο στη Βενεζουέλα που δεν ξέρουμε γιατί θα χρησιμοποιηθεί ε, με τους δικτάτορες. Και δεν ξέρουμε ε, γιατί είστε τόσο δειλοί, γιατί δεν χρησιμοποιείτε όλα τα διπλωματικά εργαλεία που έχετε στη διάθεσή σας. Η βία γίνεται όλο και περισσότερη θα πρέπει να επιβάλλεται επικυρώσεις εξατομικευμένες για κάθε δημόσιο υπάλληλο. Εγώ είδα πώς τα πρώτα χρόνια ε, αντιστάθηκαν στις κυρώσεις και όταν ήμουν φυλακισμένος κατάλαβα τι σημαίνουν αυτές οι κυρώσεις. Όταν οι δημόσιοι υπάλληλοι άρχισαν να σκέφτονται λίγο του τι κάνουν γιατί καταλαβαίνουν ότι τους παρατηρούν. Είδα αλλαγές από τις κυρώσεις στο πώς συμπεριφέρονται οι διάφοροι ε, κρατικοί λειτουργοί λόγω των κυρώσεων, γιατί οι ίδιοι θέλουν ε, τα ε, λεφτά που βγάζουν να τα χαρούν. Θέλουν οι οικογένειές τους να ζουν ελεύθερες. Οι εξατομικευμένες λοιπόν κυρώσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται, γιατί δεν υπάρχουν δικαστήρια για να δικαστούν αυτοί οι άνθρωποι οι κυρώσει, Πείτε μου εσεί, Μητέρα που είναι σε νοσοκομείο. Απελπισμένη γιατί δεν έχει φάρμακα. Τι, τι διαφορά της κάνει που έχουν παγώσει τους λογαριασμούς ενός ε, διεφθαρμένου στρατηγού. Υπάρχει κόσμος που το χειραγωγεί αυτό το επιχείρημα και λέει όχι, οι κυρώσει επηρεάζουν τον πληθυσμό. Όχι, είναι εξατογικευμένες κυρώσει που εφαρμόζονται σε διαφθαρμένους κρατικούς λειτουργούς και όχι στον τόπιο πληθυσμό το νέο ο οποίος προσπαθεί να ξεφύγει από τα σύνορα και πεθαίνει στο δρόμο του δεν τον νοιάζει καθόλου αν πάγωσαν ή όχι τους λογαριασμούς ενός διεφθαρμένου στρατηγού. Αντίθετα είναι και μια ανάσα που τους δίνεις. Ότι στο κάτω-κάτω κάποιο είδος δικαιοσύνη υπάρχει. Και ο στρατιωτικό που είναι δίπλα του, που βλέπει πω το σύντροφό του, ε, στο σύντροφό του επιβάλλανε κάποιο είδου τέτοια κύρωση, ε, θα κάνει ένα βήμα πίσω γιατί δεν θέλει να είναι ο επόμενος που θα του παγώσουν το λογαριασμό. Όπως σα είπα, θα πρέπει να του πείτε στους νέους του κόσμου ολόκληρου πως τα ε, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ε, για όσους δεν σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, είναι εσχρά και τιμωρούνται. Και γι' αυτό σας καλώ να συνεχίζουν να επιβάλλετε, να, σας, σας παροτρύνω να συνεχίζετε να επιβάλλετε κυρώσεις σε στρατιωτικούς, όχι μόνο στην Βενεζουέλα, στην Ικαραγώ, οπουδήποτε, εξατομικευμένες κυρώσεις εναντίον αυτών των ανθρώπων. Ο διάλογος δεν είναι αποτελεί εναλλακτική, ούτε στρατηγική, αλλά συνεχή ανάγκη θα πρέπει να είναι κάτι το σίγουρο. Αλλά ο διάλογος αυτός παράλληλα, εάν δεν συνοδεύεται από κάποιο είδους πίεση, θα είναι απλώς μία ανοησία. Για να είναι αποτελεσματικό ο διάλογος θα πρέπει η δικτατορία να αισθάνεται πως ο κόσμος πια δεν τους δέχεται, η ανθρωπότητα δεν τους δέχεται. Στην Ευρώπη έχουμε τους ε, παράνομους ε, πρέσβεις αυτής της δικτατορίας. Γιατί? Φανταστείτε πως έχουν έρθει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στρατιωτικοί και σας βγάζουν από τις θέσεις σας και σας φυλακίζουν. Αυτό έγινε στη Βενεζουέλα. Ο Χουάν Ρεκεσέ, που είναι βουλευτή νέο, είναι αυτή τη στιγμή κρατούμενος και βασανίζεται και είναι βουλευτή. Και οι πρέσβεις αυτών, αυτής της δικτατορίας είναι στην Ευρώπη σαν να μην τρέχει τίποτα. Και ζουν ε, με τα προνόμια των ελευθέρων χωρών όταν επιβάλλουν στον πληθυσμό τη μιζέρια και τη φτώχεια και την πείνα ο διάλογος είναι αποτελεσματικός όταν συνοδεύεται από πίεση και από μια απόκριση από την ανθρωπότητα που θα πει όπως είπατε εσείς όχι στη δικτατορία. Όχι στους δικτάτορες. Διαφορετικά θα σας κοροϊδεύουν όπως σας ε, κοροϊδεύαν από τη Δομινικανή ε, όπως ε, κοροϊδεύσαν τη Δομινικανή Δημοκρατία, όπως κοροϊδεύσαν το Βατικανό και τον Παναμά, εδώ και 20 χρόνια κοροϊδεύουν. Και το πιο ενδιαφέρον θα ήταν η καθολική δικαιοσύνη και η εφαρμογή του καθολικού δικαίου να προχωρήσει, δηλαδή σε άλλα δικαστήρια, και συνέβη αυτό, εδώ στην Ευρώπη, να δικάζονται εγκλήματα κατά ε, ε, τα εγκλήματα βασανιστήριων στην Βενεζουέλα, για παράδειγμα. Γιατί αυτοί που έχουν βασανιστεί στη Βενεζουέλα δεν είναι μόνο τα παιδιά που, πεθαίνουν ε, στη Βενεζουέλα. Ε, όπως τα παιδιά που πεινάνε στην Αφρική δεν είναι μόνο παιδιά της Αφρικής, είναι παιδιά. Και οι βασανισμένοι στη Βενεζουέλα είναι βασανισμένοι. Όταν έχουμε λοιπόν καθολική δικαιοσύνη μέσω της σύμβασης κατά των βασανιστήριων, μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αυτή τη σύμβαση για να δικάσει τους υπευθύνους για ε, βασανιστήρια που έχουν λάβει χώρα στη Βενεζουάλα σε δικαστήριο οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Θα μπορούσαμε και εδώ στην Ευρώπη. Γιατί το ε, δικαστήριο δεν κάνει βήματα, δεν θέλει να κάνει τίποτα το δικαστήριο για τα εγκλήματα ε, αυτά το γνωρίζετε κι εσείς, το γνωρίζουμε κι εμείς. Εγώ λοιπόν πιστεύω ε, στις ε, ε, κυρώσεις και στον πραγματικό διάλογο, στην πραγματική πίεση και στην εφαρμογή της καθολικής δικαιοσύνης. Που είναι η καλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια που μπορείτε να μας στείλετε και η καλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια είναι να πείτε στον Νικολάς Μαδούρο φτάνει. Και ένας τρόπος να το πείτε αυτό είναι να αφαιρέσετε τα διαπιστευτήρια αυτών των παράνομων ε, πρέσβεων που έχετε στις χώρες σας και να απαιτήσετε την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. Μία ώρα, ένα λεπτό σε ένα κελί είναι κόλαση. Είναι μια κόλαση που δεν μπορείς να την ξεχάσεις. Και δεν μπορούμε να σταματήσουμε το χρόνο. Οι άνθρωποι αυτοί είναι στις φυλακές, σε κελιά, σε παράνομες φυλακές, νέοι άνθρωποι, μεγάλοι άνθρωποι, γυναίκες που υποφέρουν. Και η πλειοψηφία των πολιτικών κρατωμένων δεν είναι καν πολιτικά πρόσωπα. Είναι πολίτες, απλοί, και τους έχουν φυλακίσει γιατί η δικτατορία χρειάζεται σε εσωτερικό επίπεδο τον πανικό και τον τρόμο για να χειραγωγεί τον πληθυσμό. Κύριε Σαλέ, πολλές ευχαριστίες. Δυστυχώς δεν έχουμε πια χρόνο, χρόνο αλλά είναι Πολύ σημαντική συζήτηση για να τη διακόψουμε στη μέση. Τρεις ερωτήσεις έχουμε ακόμα και παρακαλώ να τις ε, περιορίσετε. Και θα θέλαμε και κάποιον από την ΕΕΔ να μας κάνει μια γρήγορη δήλωση. Ιδάλλως θα σας ζητήσω να απαντήσετε πολύ γρήγορα στο τέλος. Ο λόγος τώρα στην κυρία Χάουταλα από τους Πράσινους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε που ήρθατε στις Βρυξέλλες και σε, στην Επιτροπή μας. Ήταν πολύ ζωντανέ και δυστυχώς και σο, σοκαριστικές οι μαρτυρίες των όσων έκαναν οι κυβερνήσεις σας. Οι επικρίσεις του κυρίου Οσμάν για, τη, για τους συμβασμούς που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις ίδιες τις αξίες της στη μεταναστευτική της πολιτική, χρησιμοποιώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα ως ε, ένα μέσο πίεσης στι συμφωνίε αυτέ. Αυτό έχει ακουστεί πολύ και στο Κοινοβούλιο και μα έχει διχάσει. Έχουμε ζητήσει από πολλέ χώρε τη συνεργασία του ε, γιατί ε, οι υποχρεώσει του δεν είναι μόνο να κρατάνε του μετανάστε μακριά από την Ευρώπη, αλλά να σέβονται και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό επιμένουμε. Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν πρέπει ποτέ να είναι υποκατάστατο ή ένα τρόπο να αποφύγουμε την εξέβρεση πολιτικών λύσεων σε καταστάσεις τόσο βαθέων κρίσεων όπω αυτή τη Βενεζουέλας. Σα ευχαριστούμε που ήρθατε σε εμά, κύριε Σαλέ. Και μια τελευταία κουβέντα. ω αντιπρόεδρο υπεύθυνοι για τις ε, επαφές που έχουμε και την επικοινωνία με τους πρώην βραβευθέντες με το βραβείο Ζαχάροφ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ. Ευχαριστώ για την σημερινή σας παρουσία και είμαι βέβαιη ότι η ερώτηση της κυρίας Σάντους και άλλων συναδέλφων για τη σημασία του βραβείου Ζαχάροφ είναι κάτι που τουλάχιστον για σας κύριε Οσμάν πιστεύω ότι έκανε κάποια διαφορά. Ήταν ένας τρόπος να έχετε καλύτερη προστασία Χαιρόμαστε πολύ που μιλήσαμε και με τους δυο σας. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Φαντάλεν από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία ερώτηση για τον κύριο Σμάν. Σα ευχαριστούμε για τον χρόνο που μα αφιερώσατε. Η ερώτηση που ήθελα να σα κάνω για την κατάσταση στη χώρα σα, στο Σουδάν. ακούσαμε ότι υπάρχουν ε, βίε ενέργειε, ε, διώξει, οι γυναίκε και τα παιδιά είναι τα μεγαλύτερα θύματα. Όμω, εγώ ξέρω μια ε, οργάνωση στο Σουδάν και ιδίω μια ομάδα του πληθυσμού που είναι διαρκώ θύματα δίωξη. Οι χριστιανοί συγκεκριμένα. Πρόσφατα συνάντησα την κυρία Μυρία Ιμπραήμ ε, για προσωπικούς λόγους. Ε, ζει αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες και, το και τον κύριο Πίτερ Γέσεκ, ο οποίος επέστρεψε στη χώρα του τη Δημοκρατία της Τσεχίας. Μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται με τους ε, χριστιανούς στο Σουδάν. Αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση, κύριο Σμάν. Και η δεύτερη είναι η εξής. Ήθελα κι εγώ μαζί σας να δω να έρχεται δεμένος πιστάγκωνα ο κύριος Αλμπασίρ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάκης. Δεν αρκεί κράτηση κατοίκων στο Χαρτούμ ε, ή μια τέτοια καταδίκη, γιατί δεν ξέρουμε αν έχει διαφύγει στο εξωτερικό. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να φτάσει κάποια στιγμή να δικαστεί, να φτάσει στα δικαστήρια. Θέλω να τον δω κλειδωμένο σε ένα κελί. Αλλά πώ θα γίνει αυτό. Ευχαριστούμε ο κύριο Μπένιον από την ομάδα Renew. Ευχαριστώ. Είχαμε ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στο Σουδάν τον Ιούλιο νομίζω και σε αυτήν την ε, ανταλλαγή εξέφρασα την ε, βαθιά μου επιφυλακτικότητα για το αν ή όχι οι διαδηλωτές που έφεραν την ε, συμβιβαστική αυτή λύση, την ε, διάμεση συμφωνία, τελικά έχουν διασυνδέσεις με το παλιό καθεστώς. Και μήπω απλώς ακολουθούν το δρόμο της κυβέρνηση, διότι θεωρώντας, βλέποντα βλέποντας μάλλον ποιοι είναι οι δράστες που υπέγραψαν τη συμφωνία αυτή από τη μία και από την άλλη οι διαδηλωτές, Ειλικρινά ε, γύρονται πορείε Είναι συμφωνία ή μήπω είναι κάποιο μέσο να καταστήλουμε τις διαμαρτυρίες και να επιτρέψουμε στα μέλη της προηγούμενης κυβέρνησης, του προηγούμενου καθεστώτος να ξαναπάρουν την εξουσία. Δεδομένων και των ιστορικών δεσμών με, τους, ε, με τον Τζάντζουιν και άλλους που βλέπουμε σε αυτές τις παραστηρητικές ομάδε. Είναι λοιπόν μια αυθεντική συμφωνία που θα μπορούσε να έχει διάρκεια. Ήθελα ένα σύντομο σχόλιο από αυτού. Και η ερώτηση προ τον κύριο Σαλέ. Το ερώτημα είναι τι κυρώσεις θεωρείτε ότι είναι ε, σκόπιμες και θα έπρεπε να επιβληθούν. Μιλάμε για κυρώσει που στοχεύουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Όμω εδώ έχουμε και μια κυβέρνηση που χρηματοδοτείται από την ε, ε, πόλη, στην αγο... το εμπόριο για το... του πετρελαίου. Η οικονομία τη Βενεζουέλα στηρίζεται στο πετρέλαιο και το ξέρουμε όλοι. Οπότε δεν θα είναι προς... στοχευμένα σε συγκεκριμένα πρόσωπα οι κυρώσει. Ούτως ή άλλως ε, η κυβέρνηση θα ενισχυθεί από όλο αυτό και θα μείνει στην εξουσία. Τότε θα ξαναρχίσουμε τι εμπορικέ συναλλαγέ με τη Βενεζουέλα για το πετρέλαιο. Δηλαδή, εάν κάποιο αντλεί το 90 και το 95% των ε, εσόδων του από μη προσωπικέ κυρώσει. Ε, τι θα γίνει με τι κυρώσει, τι χρησιμότητα έχουν. Ε, οι πετρελαϊκέ κυρώσει θα μπορούσαν να πλήξουν όλο τον πληθυσμό όμω. Θα έπρεπε να είμαστε πιο άμεση στι κυρώσει που επιβάλλουμε, αλλά Πού είναι η σωστή λύση. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Θα παρακαλέσω του συναδέλφους μου να είναι σύντομες τις απαντήσεις τους. Κύριος Μάνι. Uh, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάιντι Χουτάλα. Βεβαίως, ε, πάντα υπάρχει συνοχή και στις θέσεις που εκφράζονται εδώ από μέρους σας, αλλά και στην στάση αλληλεγγύη που δείχνετε προς ε, το Σουδάν. Να απαντήσω και στην ερώτηση. Ποιες είναι οι θέσεις και της παρούσας αλλά και της προηγούμενης ε, κυβέρνησης όσον αφορά την προστασία της ανεξιτρισκείας. Ο κύριος Πίτετσεκ και άλλοι Σουδανοί από την περιοχή ε, των την ορεινή περιοχή Σούμπα, οι οποίοι κατηγορούνται ότι είναι χριστιανοί, χωρίς να μπορούν να απολογηθούν. Εγώ ήμουν ένας από τους νομικούς που τους ε, υπερασπίστηκαν. Δεν υπάρχει ελευθερία θρησκείας, δεν υπάρχει στη χώρα μας δυνατότητα κανείς να εκφράσει διαφορετικές ε, θρησκευτικές πεπιθήσεις. Υπάρχει ένα είδος ρατσισμού, αραβικού ρατσισμού. Και δεν υπάρχει απολύτως καμία πολυμορφία και έκφραση άλλων θρησκευτικών ε, πεπιθήσεων και πρακτικών δεν επιτρέπονται οι θρησκευτικές τελετές και προσπαθούμε να επιτρέψουμε σε αυτές τις θρησκευτικέ ομάδες, τις άλλες θρησκείες να ε, υπάρξουν, να επιβιώσουν. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση και από μέρους της παρούσας μεταβατικής κυβέρνησης. Επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται για μια νέα κυβέρνηση, δεν πρόκειται για πολιτικούς, πρόκειται για την συνέχιση της προηγούμενης στρατιωτικής κυβέρνησης. Και πρόκειται για άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα, όπως ο πρόεδρος, ο παρόν πρόεδρος, των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και πρόκειται για άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα. Σήμερα είναι ο συγκεκριμένος αντιπρόεδρος της παρούσας μεταβατικής κυβέρνησης. μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου και μάλιστα προστατεύεται εξαιτίας και χάρη συγγνώμη, αυτής της ιδιότητάς του. Προστατεύεται δεν καλείται να απολογηθεί, να λογοδοτήσει για την σφαγή παραδείγματο χάρη της 6ης ε, Ιουνίου, αλλά και άλλες ε, βιαιότητες και σφαγές που έλαβα χώρα στην ε, περιοχή αυτή και στην πόλη της Χαρτούμ. Χρειάζεται απαραίτητα μία ανεξάρτητη ερευνητική επιτροπή, μία διεθνής Επιτροπή η οποία θα διερευνήσει όλες αυτές τις εγκληματικές πράξεις και θα πρέπει να μπορούν να προσφύγουν τα θύματα αυτών των βιωτήτων σε ένα ανεξάρτητο διεθνές ποινικό δικαστήριο. Ο Τάγκαλο, ο οποίος είναι ένας σημαντικός, μια σημαντική προσωπικότητα, επικεφαλής ε, της ε, ομάδας, η οποία σήμερα κατηγορείται και όπως ε, καταλαβαίνετε υπάρχουν παράλληλες στρατιωτικές δυνάμεις. Πρόκειται για μια κατάσταση η οποία απειλεί όχι μόνο την ασφάλεια και την ειρήνη στο Σουδάν, αλλά και τις γύρω περιοχές, την Δυτική Αφρική, τη Λιβύη. Επαναλαμβάνω, η σύνθεση αυτών των στρατιωτικών και παραστρατιωτικών δυνάμεων ουσιαστικά πρόκειται για μισθοφόρους, οι οποίοι προέρχονται από γειτονικέ χώρες και εθνότητες. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω γιατί ανέχεστε αυτήν την κυβέρνηση, τη μεταβατική κυβέρνηση, η οποία δεν είναι παρά η συνέχεια της προηγούμενης κατάστασης. Γιατί συνεργάζεστε μαζί της. Επαναλαμβάνω ότι σήμερα είναι απαραίτητο να επανέλθουμε στη δημοκρατία και να υπάρξει ανεξάρτητη δικαιοσύνη και να πάψει αυτή η ατιμορρησία που επικρατεί στη χώρα μας. Όντως, το πετρέλαιο ήταν η μεγάλη πηγή χρηματοδότησης αυτού του καθεστώτος. Και με τα δολάρια τα οποία προέρχονται από το πετρέλαιο αγοράζουν όπλα και χρηματοδοτούν όλες τις επιχειρήσεις, τις εγκληματικές επιχειρήσεις τους. Αλλά δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι και η κοκαίνη. Γιατί τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει ανάμεσα στα σύνορα Κολομβίας και Βενεζουέλας. Μη Μιλάτε εδώ για τον Αμαζόνιο και τη Βραζιλία, αλλά υπάρχει και η Βολιβία και το καταραμένο τρίγωνο μεταξύ μας, ε, γιατί εσείς μιλάτε για πολιτική εξουσία, εγώ μιλώ για εγκληματικές ε, οργανώσεις που μέσω του λαθρεμπορίου ναρκωτικών ε, χρηματοδοτούν τις δράσεις τους γιατί κάνουν λαθρεμπόριο ναρκωτικών, ε, ορυκτών, διαμαντιών, χρυσού. Οπότε χρησιμοποιούν το τρίγωνο αυτό το γεωγραφικό στην, ε, μεταξύ Βολιβίας, Κολυμβίας και ε, Βενεζουέλας ε, για να φτιάχνουν περισσότερη πάστα κοκαίνης η οποία μετά μοιράζεται στα πέρατα του κόσμου. Οπότε οποιαδήποτε δράση επιτρέψει αυτές οι δομές χρηματοδότησης να ξυλωθούν δεν είναι μόνο αποτελεσματική είναι και απολύτως απαραίτητη. Γι' αυτό είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει έναν τρόπο μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών ή κάποιου είδου σώματο να ε, κάνει επιχειρήσεις για να μειωθεί αυτή η δράση. Γιατί μπαίνουν και βγαίνουν τα ναρκωτικά στην Ευρώπη. Μπαίνει και βγαίνει στην Ευρώπη κόσμος που η δουλειά του είναι να κάνει ξέπλυμα χρημάτων. Στην Ισπανία. Εγώ ε, ζω στην Ισπανία. Οι Ισπανοί βουλευτέ το γνωρίζουν. Πώ πάνε και αγοράζουν τα πιο ακριβά κτίρια στη Μαδρίτη. Πήγα και στο Παρίσι. Και στην Ιταλία. Και είναι ε, ο τρόπος με τον οποίο κάνουν ξέπλυμα μέσω τέχνης, μέσω ε, real estate και νομίζω ότι αυτές τις επιχειρήσεις που κάνουν εξεπλήματος, οι μυστικές υπηρεσίες κάθε ε, ε, χώρας μπορούν να τις αποκαλύψουν. Δεν ξέρω, χρειάζονται κάποια κίνητρα για να το κάνουν. Πρέπει να εργαστούμε περισσότερο έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ανακρίσεις και να συλληφθούν, να ανοιχνευθούν, να συλληφθούν και να εξοδοτερωθούν αυτοί οι τρόποι χρηματοδότησης, αυτά τα logistics που χρησιμοποιεί το καθεστώς. Και όχι μόνο να δούμε τη Βενεζουέλα ως μεμονωμένο παράδειγμα, αλλά τη σχέση που έχει με τη Βολιβία, με την Ικαράγουα, με την Κούβα. Γιατί έχουμε αυτό το τρίγωνο, το τέλειο τρίγωνο, για το λαθρεμπόριο ορυκτών και ναρκωτικών. Η παραγωγή κοκαίνης είναι στα πιο υψηλά επίπεδα αυτή τη στιγμή. Και επειδή έχει μειωθεί το, η τιμή του πετρελαίου, η κοκαίνη ε, είναι πλέον ε, στο τόπ της χρηματοδότησης. Υπάρχει αυτό το καρτέλ. Και γιατί λέγεται καρτέλ του Λοσόλες, γιατί ε, το καρτέλ των ήλιων, γιατί οι, στρατηγοί στη Βενεζουέλα έχουν έναν ήλιο στο πέτο. Τη συζήτηση αυτή την έκανα με το διευθυντή του κρατηρίου εκεί που ήμουνα, ο οποίος μετά από τέσσερα χρόνια μου τα είχε πει όλα, γιατί φαντάζεστε τέσσερα χρόνια εκεί μιλάγαμε. Οι ίδιοι δικαιολογούν την αποστολή κοκαίνης στη ΣΥΠΑ και στην ε, Ευρώπη ως κομμάτι της μάχης κατά του υπεριαλισμού και κάτω από αυτή την κοροϊδία ξεπλένουν την ενοχή τους για το γεγονός ότι καταστρέφουν άρρωστους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Γιατί παράγουν και στέλνουν κοκαίνη στην Ευρώπη και στην στη ΣΥΠΑ. Και για αυτούς δεν είναι έγκλημα. Είναι μάχη. Είναι τρόπος, ένας τρόπος ακόμα να κάνουν πολιτική μάχη. Έτσι Έτσι συμβαίνει και είναι σκληρό και είναι και παράλογο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να ε, ξυλώσουμε αυτές τις επιχειρήσεις, είτε έχουν να κάνουν με εμπόριο πετρελαίου, είτε με εμπόριο ναρκωτικών. Κύριος Μαν, κύριε Σαλέου. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα μαζί σας. Είναι σημαντική μέρα γιατί σήμερα θα, θα ψηφίσουμε και για τους επόμενους ε, βραβευθε... ψηφίους για το βραβείο Ζαχάρο που πρόκειται να βραβευθούν. Ε, νομίζω ότι με την επίσκεψή σα βλέπουμε ότι έχουμε μια καλύτερη επισκόπηση των πραγμάτων, αλλά ξέρουμε ότι θα συνεχίσετε να υψώνετε και τη φωνή σα για να προασπιστείτε του υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι πολύ συγκινητικέ λοιπόν οι μαρτυρίε σα για όσα συμβαίνουν στι χώρε σα. Αλλά μα μάθατε και κάτι ιδιαίτερα πολύτιμο. Οι συστάσει ακριβώ για το τι μπορούμε εμεί να κάνουμε ω Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωκοινοβουλίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα για να σα στηρίξουμε. Το σημειώνουμε και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ladies Κυρίες και κύριοι, ζητώ συγγνώμη. Ξέρω ότι έχουμε καθυστερήσει σχεδόν ένα μισάωρο. Αλλά δεν ήθελα καθόλου να διακόψω αυτή την τόσο σημαντική συζήτηση. Θα ήθελα να προχωρήσουμε, χωρίς καθυστερήσεις, στην παρουσίαση της πρώτης έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας βάσει τη τρέχουσα νομοθεσία για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία στον κόσμο 2018. Θα δώσω αμέσω το λόγο στην κυρία Βίσλερ Λίμα από το ΕΛΚ για να μα παρουσιάσει την ε, έκθεσή τη, το σχέδιο έκθεση. Προφανώ είναι καθοριστικό τμήμα τη δουλειά μα η έκθεση αυτή. Μα επιτρέπει να συνεισφέρουμε στι δράσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να δούμε πώ εργάστηκε από αυτών των θεμάτων του 2018. Και γι' αυτό θέλουμε να διαμορφώσουμε και την σχετική δουλειά των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Συμπεριλαμβάνονται πολιτικέ συστάσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΕ και του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών. Ήθελα να σα ενημερώσω ότι η συγκέντριά μα βασίστηκε στην ετήσια έκθεση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο στι 13 Μαου φέτο. Η αγγλική εκδοχή του σχεδίου έχει ήδη ε, αποσταλεί στις 30 Σεπτεμβρίου και η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 22 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Και τώρα, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, ο λόγος στην εισηγήτρια την κυρία Βεσλέρ Λίμα ε, και την ευχαριστούμε για ό,τι έχει κάνει. Ευχαριστώ. Καταρχάς ε, να ευχαριστήσω την ομάδα. Την ομάδα που με βοήθησε να συντάξω σωστά, χωρίς λάθη και στην οριστική της μορφή αυτή, αυτό το σχέδιο έκθεσης. Στην αρχή ασχολούμαστε με το κείμενο που έχουμε από τον ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και από το Ευρωκοινοβούλιο Δεν θα περάσω σε λεπτομέρειες, διότι φαντάζομαι ότι δεν έχουμε χρόνο. Θα δούμε λίγο την δομή και μετά ίσως να κοιτάξουμε τις λεπτομέρειες εφόσον θέλετε. Οι επτά, τα επτά πρώτα σημεία αφορούν τις συστάσεις του ΟΗΕ. Με συγχωρείτε, αλλά καλύτερα να τα πω στα γαλλικά. Ευχαριστώ πολύ και με συγχωρείτε. Τα επτά πρώτα εκτιμώντα λαμβάνουν υπόψη του ε, τα διεθνή κείμενα και τι συστάσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση καθώ και τα προγράμματα δράση. Στην συνέχεια έχουμε κείμενα πιο εξειδικευμένα τα οποία αφορούν την ε, ε, άνεξη θρησκεία, την βιώσιμη ανάπτυξη, τα προγράμματα δράσης για την ισότητα των φύλων, ένα κείμενο για τη βία κατά των γυναικών και την οικογενειακή βία, τη βία κατά των παιδιών ή των ανθρώπων με αναπηρίες, για τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις εταιρείε, ε, για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες. Δύο κουκίδες μετά, δύο παύλες μάλλον, που έχουν να κάνουν με την προστασία των ε, ανθρώπων και μετά την ε, παγκόσμια στρατηγική, το Διεθνές Δικαστήριο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ε, χάρηκα πολύ που η έκθεση του 2018 πράγματι αναφέρεται στην πρωτοβουλία για τις καλέ ιστορίες σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τι θετικέ εμπειρίες. Είναι σημαντικό να μπορούμε να δώσουμε και θετικά παραδείγματα και αυτό έχει ήδη γίνει. Τα τρία επόμενα σημεία. Αναφορές στην ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο. Μετά υπάρχει αναφορά στο βραβείο Ζαχάροφ και βεβαίως στη οικονομία ε, και τη σχετική διαδικασία. Και μετά μια έκθεση προς την ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Αυτά για τα εκτιμώντας τώρα για το κύριο σώμα του, της έκθεσης. Τα δύο πρώτα υπογραμμίζουν την ε, Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αναφέρουν τη δέσμευσή μας για την ε, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Το επόμενο αφορά και πάλι την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ το Γ και το Δ αφορούν την δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης περισσότερο. Έπειτα, Υπάρχει αυτή η παρατήρηση για το γεγονός ότι γνωρίζουμε ότι η δημοκρατία μπορεί να απουσιάσει σε κάποιες στιγμές, οπότε τότε χρειάζεται κάποια δημοκρατική μετάβαση. Δηλαδή δεν είναι κάτι που γίνεται με ένα, ένα με μια κίνηση των δαχτύλων από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά χρειάζεται χρόνο. Έτσι, ε, περνάμε στα διαφορετικά σημεία για το θέμα των φύλων, τη διάσταση αυτή και στο πρώτο σημείο λέμε ότι ανησυχούμε για τις επιθέσεις που υπάρχουν κατά της δημοκρατίας. και την ε, άνοδο των αυταρχικών καθεστώτων αναφέρονται όλα σε αυτό. Δεύτερον, αναφερόμαστε στα θεμεόλη δικαιώματα τα οποία σεβόμαστε πλήρως και τη δημοκρατία και λέμε ποιες είναι οι χώρες που έχουν εγγράψει τα δικαιώματά τους αυτά στη συνταγματική τους λειτουργία και πρέπει να αγωνιστούν. Δεν πρέπει να παραμείνουμε αδρανείς ή σε παθητική στάση, αλλά πρέπει να δώσουμε τον αγώνα αυτό. Στο τρίτο σημείο στο τρίτο σημείο ε, έχουμε την κατάσταση σε σχέση με τις ένοπλες συγκρούσεις. Θάνατοι, εκτοπισμοί, η κατάσταση που βλέπουμε στις πόλεμες περιοχές. ουσιαστικά ε, αρνούμαστε την έκφραση ανθρωπιάς προς τους ε, ανθρώπους εκεί. Πρέπει να εστιάσουμε στους τόπους όπου υπάρχει πόλεμος και ένοπλες συγκρούσεις. Τέταρτο σημείο δίνει έμφαση στο γεγονό ότι υπάρχουν ε, πλήγματα κατά του πολυμερού συστήματος διπλωματεύσεων ανά τον κόσμο, ακόμα και στις χώρες όπου βλέπαμε τη δημοκρατία να υπερτερεί, να δεσπόζει. Η δημοκρατία ε, πάει χέρι, με την ε, πολυφωνία ε, σε διεθνές επίπεδο και εδώ βλέπουμε ξαφνικά μια αναδίπλωση, μια πιστοχώρηση και σε κάποιον ε, Το πολυμερές σύστημα διαπραγματεύσεων είναι πολύ σημαντικό. Το πέμπτο σημείο λέει ότι πρέπει να αντιδράσουμε. Κατά των επιθέσεων που έχουμε στα ανθρώπινα δικαιώματα, εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το επόμενο σημείο μιλάει για την αντίδραση που θα πρέπει να έχουμε για την ισότητα των φύλων, κατά της διακριτικής μεταχείρισης, κατά της βίας εις βάρος των γυναικών. Το 7 αφορά τα παιδιά, το 8 α, ανθρώπους με αναπηρίες. Και στο 9 έχουμε ένα κατάλογο που σε καμία περίπτωση δεν είναι διεξοδικός και μπορούμε να δούμε πώς θα τον συμπληρώσουμε αν χρειαστεί. Αλλά Εδώ λέμε διακριτική μεταχείριση βάσει της εθνικότητας, της θρησκείας, των πεπιθήσεων, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ηλικίας. Το διαβάζω στα αγγλικά. Έπειτα, το δέκατο σημείο αφορά τους εσωτερικούς εκτοπιστέντες και με δύο τρόπο και με μία μόνο φράση, παρόλο που είναι κάπως σύντομο, προσπαθούμε πραγματικά να αναφέρουμε τους λόγους ε, του, της ε, υποχρεωτικής αυτής εξαναγκαστικής μετακίνησης. Σας το διαβάζω για να δείτε πώς Προσπαθήσαμε έτσι πολύ συγκεκριμένα να εντοπίσουμε τους λόγους των εσωτερικών εκτοπισμών ε, υιοθετεί την άποψη ότι η πολιτική διωγμή, ο λοιμός, η εσωτερική ανασφάλεια, οι κακές συνθήκες ανάπτυξης και οι παρενέργειες των κλιματικών αλλαγών στις φτωχότερες χώρες του κόσμου, όλος ιδιαίτερος, πυροδοτούν τον ε, κίνδυνο της ε, αναζωπήρωσης ε, εχθροπραξιών συγκρούσεων και του εσωτερικού εκτοπισμού πληθυσμών. Το ενδέκατο σημείο αναφέρει το γεγονός ότι η παραπληροφόρηση είναι ένα πραγματικό πρόβλημα και θέτει ένα αμφιβόλο τη δημοκρατία. Έπειτα οι δράσεις μας. Αυτό που θα έπρεπε εμείς να κάνουμε και αναφέρονται ξανά τα άλλα σημεία. Ο τίτλος είναι «Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα να γίνει αποτελεσματικότερη». Στο 12 με 15 Ασχολούμαστε πολύ συγκεκριμένα με το θέμα αυτό. Στο 12 έχουμε ευθυγράμμιση όλων των ιστορικών πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τη διεθνή διάσταση. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, ό,τι κάνουμε στην εξωτερική μα πολιτική. Μακρηγορώ πολύ ακόμα και έτσι. Πω πω, θα προσπαθήσω να βιαστώ. Στο 13. έχουμε το εμπόριο και στο 14 βάλαμε το οποιοδήποτε πολιτικούς και οικονομικούς φραγμούς. Στο 15 υπογραμμίζουμε τις προσπάθειες που κάνει ο ειδικό απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στα επόμενα με συγχωρείτε, θα ξαναμιλήσω αγγλικά, ελπίζω ότι θα είναι πιο εύκολο έτσι. Το επόμενο τμήμα του κειμένου παρουσιάζει πιο συγκεκριμένε δράσει για να προστατεύσουμε και να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία προσπαθεί να κάνει πιο ανάγλυφα τα σημεία που ήδη αναλύσαμε. Το πρώτο σημείο είναι η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και ο χώρο που πρέπει να, στην, να δοθεί στην κοινωνία των πολιτών. Το δεύτερο, είναι μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στι ε, συγκρούσει και τι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που είναι δημοσίω γνωστέ. Στο 17 αναφέρουμε το θέμα τη ατιμορρησία και του πώ είναι σημαντικό να καταπολεμηθεί. Το είδαμε και μόλις πριν από λίγο με τους βραβευθέντες, τους νικητές του βραβείου Ζαχάροφ και μετά το 18 αναφέρει το Διεθνές, δικαστήριο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και την ανάγκη να μπορέσει ο κόσμος να έχει πρόσβαση σε παγκόσμια απόδοση δικαιοσύνης από το διεθνές σύστημα ε, ώστε να επιβληθούν σωστέ κυρώσει. Το, 19, το 19 αναφέρεται στον κατάλογο Μανίτσι και το επόμενο σημείο αναφέρει του υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο 20 μιλάμε για την ε, πολύτιμη συνεισφορά του των ακτιβιστών. Στο 21 μιλάμε για την ισότητα των φίλων. Στο 22 για τα παιδιά, τα δικαιώματα των παιδιών. Στο 23 για τα δικαιώματα των ανθρώπων με ειδικέ ανάγκες και στο 24 για την ανεξιθρησκεία και τις θρησκευτικέ πεπιθήσεις. Σχεδόν ολοκλήρωσα. Ο επόμενος τίτλος είναι οι επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε δύο εδάφια εδώ για το γεγονός ότι οι δραστηριότητες όλων των επιχειρήσεων πρέπει να συμφωνούν απολύτω με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αναφέρεται στις κατευθύνες γραμμές του ΟΗΕ για τις εταιρείε και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 26η παράγραφος σημειώνει ότι είναι θετικό το σύστημα των GSP ε, των γενικών δασμολογικών προτιμήσεων και εδώ ε, έχουμε τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα από τι ψευδεί ειδήσει, την παραπληροφόρηση και τι μαζικέ υποκλοπέ και παρακολουθήσει. Η επόμενη παράγραφο αφορά του πρόσφυγε και μετανάστε και ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τα γενεσιουργά, γενεσιουργά αίτια τη μετανάστευση και των μεταναστευτικών ρόλων παγκοσμίω. Αναφερόμαστε και στην ατζέντα του ΟΗΕ για το 2030. Η επόμενη παράγραφος αφορά την έκθεση του ΟΕ και λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να προωθεί τον εκδημοκρατισμό και τις διαδικασίες για να υπάρξει ευρωπαϊκή συμμετοχή στα ανατολικά και νότια της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να επιδιώξουμε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών. Η τριακοστή και τελευταία παράγραφος έχει να κάνει με τη σταθερή στήριξη στις δημοκρατικές διαδικασίες. Με συγχωρείτε, δεν μπορούσα να συντομεύσω περισσότερο. <laughs> Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ήθελα να σας πιέσω, αλλά είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε και τους συναδέλφους. Η Σκιώδης, καταρχήν, εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Θα είμαι πολύ σύντομος. Τα περισσότερα σημεία τα ανέφερε ήδη η συγκήτρια, θα συνεργαστούν. Πριν μπω όμως στις λεπτομέρειες, να πω ότι και φέτος, δυστυχώς, η ετήσια έκθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα εγκριθεί σχεδόν με μια καθυστερήση διετίας. Αυτό υπονομεύει την αξιοπιστία του ίδιου του Κοινοβουλίου και εν μέρη η καθυστέρηση οφείλεται στις ευρωεκλογέ, εν μέρη στους διαδικασίες που είναι πολύ χρονοβόρες και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο το ίδιο. Εδώ λοιπόν ίσως θα μπορούσα να επαναλάβω την πρόσκλησή μου προς την Υποεπιτροπή Ντρουά και να πω ότι καλό θα ήταν να έχουμε διαθεσμικό διάλογο με την ΕΕ και το Συμβούλιο. Στη επόμενη ετήσια έκθεση να εγκριθεί τουλάχιστον στο πρώτο εξάμεινο της επόμενης χρονιάς και να ανακτήσουμε την αξιοπιστία που θέλουμε να έχει αυτή η έκθεση. Αυτή. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του σχεδίου έκθεσης, θεωρώ ότι είναι πολύ καλή η αφετηρία καλύπτεται μια ποικιλία επιχειρημάτων όπως μας παρουσίασε μόλις η εισηγήτρια ε, και κυρίως ε, με χαροποιεί ιδιαίτερα η συγκεκριμένη αναφορά των ε, ρητρών διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εμπορικέ συμφωνίες και υπάρχει και η ομάδα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είχε οργανωθεί από την υποεπιτροπή μας πέρσι. Θα θέλαμε να δοθεί μόνιμο τέρμα τη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και εδώ, σε αυτό το τελευταίο σημείο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω η Επιτροπή μα, πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση και να προωθήσουν ένα πραγματικό εργαλείο τη Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη ατιμορρησία. Και παρόλο που χρειάζεται μια έκθεση συνοπτική, υπάρχουν ακόμη περισσότερα θέματα ε, για τα οποία θα υποβάλω τροπολογίε και τα οποία θα θέλουν να συμπληρωθούν. Συγκεκριμένα τα δικαιώματα των ΛΟΑΔ, συγκεκριμένα τα δικαιώματα όσων μεταναστών δεν εντάσσονται παρκώς σε διάφορα συστήματα στον κόσμο. Και μετά η λυπής προβολή που δίνουμε στο θέμα αυτό. Επίσης θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τις μνήες στην ε, μεταναστευτική πίεση, κάτι που κάνει η ίδια η συγγήτρια ούτως ή άλλως, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για μια πραγματική πρόκληση των καιρών μας Γι' αυτό και τα υπόλοιπα θέματα θα ε, ε, συντάξω τροπολογίε και θα τι υποβάλω εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Υποσχέθηκα να είμαι συνοπτικό και κλείνω τώρα. Η έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι μόνο ένα από τα σημαντικότερα κείμενα που έχουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εκπροσωπεί και μια σημαντική ευκαιρία να αποστείλουμε ένα σαφέ ηχηρό μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προ τον υπόλοιπο κόσμο. Ένωση που θα πρέπει να αναλάβει πρωταγωνιστικότερο ρόλο, χρησιμοποιώντα όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή τη, για να βεβαιωθεί ότι είναι, έχουν πρωτοκαθεδρία τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προστατεύουμε σε οποιοδήποτε διάλογο, επικοινωνία, συνομιλίε έχουμε στην εμπορική μα πολιτική, σε αυτέ για τη διεύρυνση, στι μεγάλε προκλήσει τη νέα εποχή. Θα πρέπει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε και μια νέα ταυτότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να την προβάλλουμε ω κάτι καινούριο και να ενισχύσουμε το ρόλο τη ώστε η παρουσία τη ε, παγκοσμίω να είναι ε, ισχυρότερη και περισσότερο στοχευμένη από ό,τι στο παρελθόν. Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Βεζολίνο, αλλά δεν βλέπω τον κύριο Γκέρενς. Ποιος θα ήθελε να πάρει το λόγο? Η κυρία Νόμενα από την <coughs> ομάδα των Πρασίνων. Ευχαριστώ καταρχήν. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω το ΕΛΚ και την Ιζαμπέλ ιδιαίτερα για αυτήν την πρόταση ψηφίσματος. Θέλω να απαντήσω σε αυτά τα σχόλια που έκανε ο κ. Παζολίνο. Ελπίζω να βρούμε λύση την επόμενη χρονιά. Εμείς σαν πράσινοι πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή βάση για να προχωρήσουμε στις τελικές προτάσεις και χαιρόμαστε γιατί κάποιες από τις ιδέες που είχαμε υποβάλει έχουν ληφθεί υπόψη. Έχουμε υποβάλει αριθμό τροπολογιών, αυτό νομίζω δεν θα σε εκπλήσει, ιδιαίτερα για θέματα που αφορούν την πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το σχέδιο δράσης, τον ειδικό απεσταλμένο για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τις δράσεις που στοχεύουν στην πρόθεση και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θεματικές ενότητες επίσης προτείνονται θέματα που αφορούν τους υπερασπιστές δικαιωμάτων του περιβάλλοντος, τα δικαιώματα των αυτοχθόνων, αλλά και το θέμα της εποπτείας, της παρατήρησης όσον αφορά την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προσβλέπουμε στη συζήτηση που θα ακολουθήσει και ελπίζουμε ότι θα συμπεριληφθούν και οργανώσεις που προέρχονται από την κοινωνία των πολιτών γιατί πραγματικά θέλουμε να ακουστούν και οι δικές τους προτάσεις. Ε, ξέρω ότι υπάρχουν διάφορες διαδικασίες που εξελίσσονται παράλληλα. Είναι πολύ σημαντικό να φτάσουμε σε ένα τελικό κύμα που θα αντικατοπτρίσει απόψε όλους, αλλά ήδη σας ευχαριστώ πολύ για την παρούσα σας πρόταση. Ποιος ε, θέλει να πάρει το λόγο εκ μέρους του ECR? Δεν βλέπω κανέναν. Ούτε ο κύριος Κράσκιν είναι εδώ. Η Γκουε. Ωραία. Εντάξει. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. ID. Όχι. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο εκ μέρους των ε, παρόντων μελών στην αίθουσα. Θα δώσω το λόγο στην ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, η κυρία Βρέτσερ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές για αυτή την τόσο χρήσιμη γνωμοδότηση και να σχολιάσω κάποια στοιχεία από αυτά τα οποία αναφέρετε και να απαντήσω και σε κάποιες από τις ερωτήσεις που μας έχετε θέσει. Η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο βασίζεται στην ετήσια έκθεση την οποία ε, υιοθετεί το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Τώρα για τη χρονική στιγμή της έγκρισης, ο κύριος Κοτσολίνο αναφέρθηκε στην έγκριση που δόθηκε με δύο χρόνια καθυστέρησης εμείς. Ε, πρέπει να πω ότι είμαστε ικανοποιημένοι γιατί βλέπουμε ότι στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις 13 Μαΐου η κατάσταση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Για την επόμενη λοιπόν χρονιά είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τις ε, ίδιες δομές και παράλληλα θα προσπαθήσουμε η έκθεση αυτή μέχρι την άνοιξη του 2020 να έχει εγκριθεί. Για τα διάφορα σημεία τα οποία έχετε θίξει στην έκθεση, και επίσης για τα όσα έχουν τονιστεί από τα μέλη τα οποία ζήτησαν το λόγο να σας πω πως εμείς όντως στηρίζουμε ε, την έκκληση αυτή για την ε, ένταξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάθε πολιτική όπως επίσης και για την έκκληση τα ανθρώπινα δικαιώματα να συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο ως θέμα συζήτηση ε, με τους εταίρους μας στις τρίτες χώρες στα πλαίσια ε, του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά σε όλο τη συνεργασία που έχουμε είτε είναι εμπορικό διάλογος είτε πολιτικός είτε κάποιο άλλο είδους διάλογος. Για την ατιμορρησία και για το Διεθνές ε, δικαστήριο, ποινικό δικαστήριο, θα ήθελα να πω πως το δικαστήριο αυτό αποτελεί ακρογωνιαία λίθο του Παγκοσμίου Συστήματος Διεθνούς Δικαιοσύνης εμείς ε, για την ε, διεύρυνση του καθεστώτος της Ρώμης εμείς κάνουμε συνέχεια βήματα και σε διμερείς συζητήσεις με, τα, με τρίτες χώρες αλλά και στα πλαίσια ευρύτερων ε, συνθήκων ε, συζητάμε το θέμα αυτό και εντάσσουμε ρήτρε σχετικές με το δικαστήριο. Επίση, θα γνωρίζετε κι εσεί πω η εντολή ε, για το νέο Καθεστώ για τα, ανθρωπίνα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα λαμβάνει περισσότερο υπόψη τα θέματα του δικαστηρίου και των αποφάσεών του σε θέματα ανθρωπίνου δικαστηρίου. Τώρα για όσου υπερασπίζονται τα δημοκρατικά και ανθρώπινα δικαιώματα συζητήθηκε εκτενέστατα και είπαμε να δούμε τη χορήγηση θεωρήσεων για παράδειγμα είναι κατευθυντήριε γραμμέ για όσου υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα έγγραφο το οποίο είναι ε, προσβάσιμο ε, και έχουμε πει πως μπορούμε να προσφέρουμε άλλωστε και προσωρινό καταφύγιο στα κράτη-μέλη ως ένα από τα προσωρινά μέτρα τα οποία εγκρίνουμε για τους ε, όσους υπερασπίζονται ανθρώπινα δικαιώματα και αυτά στα πλαίσια των προσπαθειών μπορούν να κάνουν οι χώρες μας ξεχωριστά. Για τα δικαιώματα του παιδιού ε, Ακολουθώ την δομή ε, των όσων μας είπε ο εισηγητής και εκεί έγιναν συγκεκριμένες, ε, συγκεκριμένες αναφορές στη διοργάνωση μιας διάσκεψης για τα δικαιώματα των παιδιών σε τροτά περιβάλλοντα. Είμαστε ανοιχτοί στο να συζητήσουμε τις δυνατότητες αυτές και πιο λεπτομερώς με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως επίσης και με τους συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα χρειαστεί να καταλάβουμε ε, ποιο είναι το πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, αλλά παράλληλα θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως γίνονται συζητήσεις για τα δικαιώματα του παιδιού και σε πολυμερή ε, βήματα και θα γίνει μια ημερήσια συζήτηση στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά από πρωτοβουλίο το οποίο ανελήφθη στην Τρίτη Επιτροπή της Νέας Υόρκης. Φέτος έχουμε ε, συζητήσει το να παρουσιάσουμε ε, το θέμα αυτό στα πλαίσια των δικαιωμάτων των παιδιών που δεν έχουν γονική ε, φροντίδα και θα πρέπει να δούμε πώς όλα αυτά θα συμπληρώσουν ε, τις ε, διάφορες πρωτοβουλίες που τρέχουν. Για την ε, θρησκευτική ελευθερία αναφέρεστε σε μία πλατφόρμα που θα επιτρέψει και στην κοινωνία των πολιτών και στους θρησκευτικού ηγέτες να έρχονται σε επαφή και θα σας υπενθυμίσω πως έχουμε την σχετική διάσκεψη και την πρωτοβουλία το, την οποία 6 Σεπτεμβρίου εκκίνησε η ύπατη εκπρόσωπος κυρία Μογκερίνη. Έτσι νομίζω έχουμε ανταποκριθεί σε αυτό το αίτημα. Και έχουμε και τη διαδικασία της Κωνσταντινούπολης και την επόμενη ε, εκδήλωση θα την κάνουμε ε, το Νοέμβριο. Για τη νέα τεχνολογία και τα ανθρώπινα ε, δικαιώματα, τώρα μιλάμε για την περισσότερη προσοχή που θα δοθεί στις αναδυόμενες προκλήσεις, όπως επίσης και στις αναδυόμενες ευκαιρίες που θα βρεθούν μπροστά μας έτσι ώστε να εξετάσουμε με ιδιαίτερη προσοχή αυτό το χώρο ε, προετοιμάζοντας το καινούριο σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία που επίσης αναφέρθηκε από την κυρία Νόημαν. Για την κυρία Νόημαν και τα όσα είπε για τους αυτόχθονες και το περιβάλλον, Στην έκθεση αναφέρθηκε πως πέρσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πρώτη φορά οργάνωσε μία εβδομάδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα για την επέτειο της ε, διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό ε, ε, διάστηκε με το φόρουμ για τις ΜΚΟ που έφερε κοντά εκπροσώπους τη κοινωνίας των πολιτών από όλο τον κόσμο και φέτος θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο για το περιβάλλον και τους όσους υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το συζητήσαμε και βασιζόμαστε και στη δική σας συμμετοχή. Εκεί λοιπόν έχουμε εστιάσει τη δραστηριότητά μας είναι ένα θέμα αναδυόμενο και κυρίως όταν μιλάμε για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι δύσκολο. Δύσκολο το θέμα και αυτοί οι οποίοι ε, κινδυνεύουν περισσότερο είναι αυτοί που ασχολούνται με το θέμα ε, της υπεράσπισης του περιβάλλοντος και της κλοπής γεών. Να σας πω πως είμαστε πάντα διαθέσιμοι για οποιαδήποτε ανταλλαγή θέλετε να κάνουμε και θέλουμε να ευχηθούμε και εμείς πως η έκθεση θα εγκριθεί ε, την κατάλληλη χρονική στιγμή στην ώρα της του χρόνου. Έχουμε εδώ εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εάν όχι, η κυρία Βίσλερ για να κλείσει το θέμα. Θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω όλους για όλες τις, όλη τη συνεισφορά στην έκθεση. Προς το παρόν ε, το σχέδιο αυτό κειμένου αποτελεί απλώς το πλαίσιο, αν θέλετε, μέσα στο οποίο θα συμπληρωθούν όλες οι ιδέες τις οποίες ακούσαμε από όλου σας. Και θα είναι πολύ μεγαλύτερο το κείμενο, πολύ πιο πολύ σέλιδο. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν όλους και είμαι σίγουρη ότι η δουλειά που θα ακολουθήσει θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για όλους. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν τόσο σύντομοι. Καταφέραμε να ολοκληρώσουμε ακριβώς στην ώρα μας. Ευχαριστώ πολύ όλους για την προσοχή σας, την παρουσία σας για αυτήν την πάρα πολύ συγκινητική και χρήσιμη συνεδρίαση. Θα ακολουθήσει και κλεισμένων το θυρών η συνεδρίαση των συντονιστών.